Dear colleagues, may I ask you to take seat? I would like to warmly welcome uh, all the... Παρακαλώ, καθίστε. Συνάδελφοι, καλωσορίζω όλους τους εκπροσώπους από τα κοινοβούλια. Σας ευχαριστώ που ήρθατε για την ανταλλαγή αυτή απόψεων για τον κύκλο του 2016 του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η στιγμή είναι κέρια για μια συζήτηση η οποία ε, βεβαίως ε, κανονικά αναφέρεται στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αλλά έχει και μεγάλη σημασία για την προετοιμασία του 2017. Λοιπόν, το κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο λαμβάνει αποφάσεις ε, στο πλαίσιο του προπολογισμού του που μπορεί να επηρεάσουν άλλα κράτη-μέλη. Σημαντικό είναι άρα να γίνει αυτή η συζήτηση που αφορά το αποτέλεσμα του κύκλου του 2015, ε, την τρέχουσα περίοδο και βεβαίως την επόμενη. Και όπως ε, ξέρετε αυτή τη στιγμή οριστικοποιείται η σχετική έκθεση, η συγητής είναι ο κύριος Σαντ και στόχος είναι ακριβώς να συνεισφέρουμε στην έκθεση αυτή πριν εγκριθεί επισήμως η ε, έκθεση. Έχει κλείσει βεβαίως η προθεσμία για τροπολογίες, αλλά πρέπει να προετοιμαστούν οι συμβιβαστικές τροπολογίες. Είναι κρίσιμη λοιπόν η στιγμή, οπότε ε, έχει μεγάλη σημασία η συνεισφορά σας. Και σε γενικές γραμμές η συζήτηση αυτή νομίζω είναι σημαντική για να δούμε τις απόψεις μας για τις μακροοικονομικές προοπτικές και επίσης τις συστάσεις που σχετίζονται ιδιαίτερα με την συνολική φορολογική στάση της Ευρωζώνης ε, και το τι θα παρουσιάσει η Κομισιόν για το 2017. Να σας μεθυμίσω ότι λόγω των πολλών παρισταμένων και για να διευκολύνουμε την συμμετοχή όλων των Εθνικών Κοινοβουλίων μόνο ένας ε, βουλευτής από κάθε χώρα θα λάβει το λόγο στον πρώτο γύρο. Βεβαίως θα προσπαθήσουμε στους επόμενους γύρους να δώσουμε τον λόγο. Έχουμε λοιπόν 20 γλώσσες σήμερα. Χρησιμοποιούμε τις κάρτες αυτές ε, για να ζητήσετε τον λόγο. Τα δίνετε στους κλητήρες. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Σάντ, για να παρουσιάσει την έκθεσή του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους βουλευτές που είναι εδώ πέρα σήμερα για την ετήσια αυτή ανταλλαγή απόψεων για τον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Για πέμπτο συνεχόμενο έτος έχουμε ανταλλαγή με τα Εθνικά Κοινοβουλία για το 2016-2017 στο πλαίσιο μιας συνεδρίασης τη Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με το τρέχον σύστημα, προσκαλούνται τα εθνικά κοινοβούλια και εξετάζουν τι συστάσεις αναχώρα τι οποίε μεταφράζουν στο εθνικό τους επίπεδο. Υπάρχουν λοιπόν τρεις φάσεις οποίε μπορούν να εμπλακούν τα εθνικά κοινοβούλια. Πρώτα απ' όλα στην ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη. Δεύτερον, όταν οι εθνικέ κυβερνήσει προετοιμάζουν τα σχέδια μεταρρυθμίσεων και σταθερότητας και τρίτον όσον αφορά τις συστάσεις αναχώρα. Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν είναι πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ή καλύτερα πώς μπορούν τα Εθνικά Κοινοβούλια να παίξουν έναν πιο ουσιαστικό ρόλο στην σύνταξη των εκθέσεων στο Εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πώς ε, βεβαίως μετά θα μπορούν να παρουσιάσουν τις εκθέσεις αυτές αφού έχουν συμφωνήσει από αυτόν σαν δικές τους. Βεβαίως είναι σημαντικό γιατί τα εθνικά κοινοβούλια ε, υπερασπίζονται το εθνικό συμφέρον και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ευρωπαϊκό θα έλεγε κανείς. Οπότε αυτό το οποίο έχει νόημα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ε, μπορεί όταν εφαρμόζεται στο εθνικό επίπεδο να μοιάζει με δηλητήριο. Βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα βεβαίω όλοι νεκροί είμαστε και βραχυπρόθεσμα όλοι κινδυνεύουμε να χάσουμε τι εκλογέ. Όμω υπηρετούμε του ίδιου ανθρώπου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε υπό το πρίσμα του πώς οι ανά χώρα εφαρμόζονται από τι κυβερνήσει. Με βάση λοιπόν τις ε, συστάσεις της ε, Κομισιόν, το ποσοστό αυτών που εφαρμόζονται έχει μειωθεί στο μισό στους προπολογισμούς 2012-2015. Ενώ οι αυτές οι οποίες δεν σημειώνεται καμία πρόοδος έχει πάει από το 30% στο 50% από το 2012 στο 2015. Βεβαίω, οι συστάσεις αναχώρα της Κομισιόν το 2016 ήταν λιγότερες σε αριθμό, ήταν πιο εστιασμένες για να επικεντρωθούν στις επίγουσες ε, ανάγκες της κάθε χώρας και βεβαίω για να τις αγκαλιάσουν περισσότερο οι χώρες. Όμως εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της ε, ασθενού εφαρμογή των συστάσεων αναχώρα και ω αποτέλεσμα αυτού σοβαρό πρόβλημα του οικονομικού συντονισμού είναι ότι δεν λειτουργεί. Υπάρχει όμως και ένα πιο θεμελιώδες δίλημα. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα σταυροδρόμι σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που από ό,τι φαίνεται πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, δημοσιονομικής πειθαρχία και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για να δημιουργήσουμε περισσότερες επενδύσεις. Ένα από τα τρία ή δύο από τα τρία ή τρία από τα τρία αλλά οπωσδήποτε το καθένα με τις δόσεις του και βεβαίως συμφωνούμε. Τις περισσότερες φορές οι διαφωνίες είναι περισσότερο δογματικές και οφείλονται σε πιστεύω, δεν θέλω να πω, προκαταλήψεις. Και φαίνεται ότι έχουμε πάει περίπου στην ε, Ενωμένη Ευρώπη του Μεσαίωνα, όπου είχαμε κυρίως θεολογικές διαφορές μεταξύ Δομινικανών και Φραγκισκανών ε, στα πανεπιστήμια της Μπολόνιας ε, Τη ορβόνη και τη Οξφόρδης. Λοιπόν, θα πρέπει όμως να βρούμε τον τρόπο για να επανέλθει η οικονομική ανάπτυξη. Σε ποιο βαθμό θα πρέπει να μειωθεί η ευελιξία και για ποιον θα πρέπει να ισχύει. Μόνο σε αυτού που είναι πολύ μεγάλοι για να χρεοκοπήσουν ή για όλους ή σε κανέναν. Επίση, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στην αγορά εργασία. Αρκούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, και οι προπολογισμοί, πως χρειάζεται κάτι άλλο για να προωθήσουμε τις επενδύσεις. Θα πρέπει να είναι μόνο δημόσιες επενδύσεις ή θα πρέπει να βρεθεί και άλλος τρόπος. Τι θα γίνει ε, σε σχέση με την ανάγκη να μην παραβιαστεί το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης ε, σε όλα αυτά. Βεβαίω θα πρέπει να αναστραφεί και ο οικονομικός μάρισμός της Ένωσης για να υπάρξει και περισσότερη οικονομική και κοινωνική συνοχή. Και βεβαίως ε, μιλώντας ε, με την εμπειρία των συστάσεων αναχώρα, τις οποίες προετοιμάζουμε, προσπαθούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Κομισιόν, εστιάζοντας σε λίγα θέματα, αντί να κάνουμε μεγάλες δηλώσεις. Προσπαθούμε να επικεντρωθούμε στο θέμα των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένων των συνθήκων του πώς καθορίζονται οι πολιτικές στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποιες συστάσεις μπορούμε καλύτερα να κάνουμε ποια συνένεση ή τουλάχιστον κάποια συμφωνία μπορούμε να περιμένουμε για το πώς θα προσελκύσουμε επενδύσεις και βεβαίως θα πρέπει να έχει η εκθεσή μας και νόημα για τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών που θα ήθελαν ακριβώς να έχουμε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη από ό,τι τα τελευταία χρόνια. Είμαι σίγουρο λοιπόν πω αυτά τα οποία θα ακούσουμε σε αυτή την συνεδρίαση θα μας βοηθήσουν πολύ σε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, ευχαριστώ πολύ Το ενισχύτη. Δεν βλέπω αν ο κύριος Φέρμπερ για το ECR. Πάμε στους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο, ο Μπαϊρακτάροφ από την Βουλγαρία. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να εκφράσω την ε, άποψη ε, της χώρας μου όσον αφορά τις ειδικές συστάσεις. Πρώτα απ' όλα να πω ότι, το, ότι η Βουλγαρία θεωρεί ότι για το 2016 είχαμε ένα προπολογισμό που λειτουργούσε πολύ καλά και ήταν εξαιρετικά ισορροπημένος. Γι' αυτό χαιρόμαστε για την ε, ιδιαίτερα θετική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, με τον τρόπο αυτό ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα σωστό, μια σωστή πολιτική διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν ε, μας αρέσει η προσέγγιση της Κομισιόν. Πιστεύουμε ότι οι συστάσεις θα πρέπει να είναι ολιγάριθμες και πιο επικεντρωμένες, πιο εστιασμένες. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε ότι υπάρχουν και στοιχεία τα οποία μπορούν περαιτέρω να βελτιωθούν έτσι ώστε να υπάρξουν καλύτερες ε, δεσμεύσεις ε, και σε τεχνικό και σε πολιτικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει ε, πραγματικά να τίνει ευήκονους στα συγκεκριμένα επιχειρήματα των κρατών μελών. Θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των διαφόρων μονάδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς επίσης και των διαφόρων επιτροπών του Συμβουλίου γιατί υπάρχουν αποφάσεις που λαμβάνονται από μία μονάδα και οι οποίες ενδεχομένως έχουν επίπτωση σε αποφάσεις της άλλης μονάδας. Ε, επίσης, ε, πρέπει να πω ότι διαπιστώνουμε ότι πολλές φορές υπάρχει έλλειψη συντονισμού, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα για την Βουλγαρία όσον αφορά η, την σύσταση 3, η οποία ε, σχετίζεται με το σύστημα ελάχιστων αμοιβών. Θα πρέπει να το δούμε μαζί με την ε, ειδική σύσταση υπαριθμών 1, η οποία αναφέρεται στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων. Επανειλημμένα η Βουλγαρία έχει πει ότι συμφωνεί με τις συστάσεις αυτές. Δεν έχουμε, ε, ε, έχουμε μάλιστα και κάποια δήλωση η οποία διαβάστηκε στην Εκοφίνα τον ε, Ιούνιο και έχουμε πει ότι συμφωνούμε με αυτές τις συστάσεις. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να αυξηθεί η βιωσιμότητα των εξειδικευμένων συστάσεων. Υπάρχουν πολύ συχνά τροποποιήσεις ε, των ε, πολιτικών ε, και σε πολλές περιπτώσεις αυτό προκαλεί αποσυντονισμό και έλλειψη εστίασης Τη όλη ε, διαδικασία. Ε, πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να ε, προσεχτεί ιδιαίτερα το σημείο αυτό. Θα πρέπει να δούμε ότι μερικέ φορέ α πούμε, διαβάζοντα τι συστάσει, βλέπουμε ότι πότε γίνεται εστίαση στην κοινωνική διάσταση, πότε στην οικονομική κτλ. Το σημαντικό για μα είναι η υλοποίηση. Θα πρέπει βεβαίω οι χώρε να είναι συγκρίσιμε, κυρίω όταν μιλάμε για διαδικασίε μακροοικονομική ισορροπία. Ε, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να ανταλλάσσουμε απόψεις και με τις άλλες χώρες. Όσον αφορά τώρα ε, τις ε, προτάσεις της ΕΚΟΝ για το ευρωπαϊκό εξάμεινο, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερως υπόψη. Θα πρέπει να ληφθεί επίγουσα δράση όσον αφορά το, το θέμα αυτό και πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να ενταχθεί και σε στρατηγική 2020 ε, οι συστάσει ε, για τη χώρα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και, ε, να συμπεριλαμβάνονται και το θέμα αυτό. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί η δράση έτσι ώστε να αρθούν τα ρυθμιστικά προσκόμματα τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν. Η βουλγαρική κυβέρνηση έχει ταυτοποιήσει 10 προβληματικά πεδία τα οποία θα ήθελε να συζητήσει περαιτέρω και για τα οποία και συγκεκριμένες προτάσεις και μέτρα έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα προσκόμματα και οι δυσκολίες αυτές. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει συνοχή και συντονισμένη δράση μεταξύ των κρατών μερών γιατί ε, οι οικονομίες των χωρών μας είναι διασυνδεδεμένες. Αν θέλουμε να επιτύχουμε αυτά αποτελέσματα θα πρέπει να έχουμε συντονισμένες πολιτικές, ε, οπωσδήποτε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και ενισχυμένο διάλογο έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα ε, προβλήματα και για να επιτύχουμε βεβαίω ε, και την ενιαία αγορά. Αλλά πιστεύω ότι η κύρια λέξη κλειδί είναι η λέξη εμπιστοσύνη. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Charles Mannion από τη Μάλτα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αναφέρθηκαν πολλά και σημαντικά στοιχεία. Κατά την άποψή μου το σημαντικότερο είναι οι επενδύσεις ή αν θέλετε η έλλειψη παραγωγικών επενδύσεων. Πρόσφατα ο κύριος Ντράγκη επιβεβαίωσε ότι η ποσοτική χαλάρωση δεν είναι αρκετά ελκυστική για να αναπτυχθούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και για να δημιουργηθούν οι απαραίτητες θέσεις απασχόλησης. Άρα δηλαδή τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να εισάγουν κίνητρα που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις. Το ερώτημα που τίθεται αυτή τη στιγμή είναι τι είδους επενδύσεις. Μιλάμε για δημόσιες ή για ιδιωτικές επενδύσεις. Κατά τη δική μου άποψη είναι απαραίτητο να υπάρχουν και δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Και πάλι λοιπόν όσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις το θέμα το οποίο τίθεται είναι το θέμα της ευελιξίας. Ευελιξία στο πλαίσιο του πακέτου δημοσιονομικής σταθερότητας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται τώρα πλέον εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και δεν έχει ληφθεί καμία αποτελεσματική απόφαση. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι ευθύνη των εθνικών κοινοβουλίων τα οποία πρέπει να επιτρέπουν κάποια ευελιξία μέσα στις παραμέτρους του Συμφώνου Σταθερότητας. Είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητο οι εθνικές κυβερνήσεις να ενθαρρύνουν πολιτικές οι οποίες στηρίζουν τις δημόσιες επενδύσεις γιατί με τον τρόπο αυτό στηρίζονται και οι ιδιωτικές επενδύσεις ή αν θέλετε να υπάρχει ένα μείγμα ε, ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, ένα είδος ΣΔΙΤ. Ε, αυτή τη στιγμή πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα πώς ε, μπορούν να ενθαρρύνουν ε, περαιτέρω τις επενδύσεις οι οποίες πάλι θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Νομίζω ότι σε αυτό το κοινοβούλιο, σε αυτό το φόρουμ, οφείλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας. Γιατί από τη στιγμή που θα ξεπεράσουμε το θέμα των επενδύσεων και των δημόσιων και των ιδιωτικών αυτομάτως ε, θα δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και αυτό θα προάγει την καλύτερη συνεννόηση ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης θα προάγει και τη στήριξη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα ανακοινωθέν σχετικά με την ευελιξία για την προσαρμογή των δομών και επιπλέον το Συμβούλιο επικύρωσε αυτή την απόφαση αλλά ε, προβλέπεται και η κεφαλοποίηση ενός έτους, δηλαδή μπορεί κανείς να επωφεληθεί από αυτές τις επενδύσεις, αλλά μόνο για ένα χρόνο ε, και δημιουργούνται ε, κάποιες αμφιβολίες, γιατί όλα αυτά είναι θέματα που δεν μπορούν να επιληθούν μέσα σε ένα χρόνο. Επόμενος ομιλητής, Αν Μούλντερ από την Ολλανδία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι οικονομίες των κρατών μελών είναι διασυνδεδεμένες και οι αρνητικές εξελίξεις σε ένα κράτος μέλος ε, μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για άλλα κράτη-μέλη. Εάν δείτε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο σύνολό της, βλέπετε ότι έπεσε τα τελευταία 15 χρόνια. Εάν ε, ακούσετε όσα λέει ο κύριος Ντράγκη της Κεντρικής Τραπεζάς, ζητάει μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη για να διατηρηθεί το ευρώ και η ευρωζώνη στάθερη. Και για να λυθούν αυτά τα προβλήματα έχουμε τις συστάσεις αναχώρα. Αυτές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν, αλλά όταν φτάνουμε στην εφαρμογή ξεκινάνε τα προβλήματα. Ούτε οι μισές από τις συστάσεις δεν εφαρμόζονται. Και το ερώτημά μου είναι τι θα κάνουμε ως βουλευτές και ευρωβουλευτές ε, και κομισιόν για την έλλειψη εφαρμογής αυτών των συστάσεων. Ποια μέτρα μπορούμε να λάβουμε, ε, πως χρειάζονται πρόστιμα ή άλλες, άλλα μέτρα. Αναμένω απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, όχι γιατί μου αρέσουν τα μέτρα ή τα πρόστιμα, αλλά επειδή θέλω μια ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα σταθερό ευρώ, έτσι ώστε οι λαοί μας να προοδεύσουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που θέσατε το θέμα αυτό, το κρίσιμο πράγματι. Η Κομισιόν κάνει κάποιες αξιολογήσεις. Ε, Παραδείγματο χάρη στην Ολλανδία έγιναν τρεις ε, ε, συστάσεις για την δύο περιορισμένη πρόοδο, στην μία έγινε υπήρξε κάποια πρόοδος. Οπότε το θέμα είναι πραγματικά για εμάς αλλά και για εσάς τα εθνικά κοινοβούλια πώς ε, αντιδράτε όταν ε, δεν τα εφαρμόζει η κυβέρνησή σας. Κοιτάξτε, εμείς παίρνουμε πολύ σοβαρά αυτές τις ε, συστάσεις. Φέτος είχαμε αυτές τις τρεις συστάσεις για την αγορά εργασίας, για τα δημόσια οικονομικά και τα συζητήσαμε στο Κοινοβούλιο. Έχουμε εκλογές του χρόνου και αυτά τα θέματα θα μας απασχολήσουν. Οπότε έχουμε τη συζήτηση στο κοινοβουλίο μας, αλλά κοιτάμε και τι γίνεται και σε άλλα κοινοβουλία. Στη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία. Ελπίζουμε και αυτοί να μεταρρυθμίσουν την οικονομία τους για να αυξηθεί η ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ειδικά οι μεγάλες χώρες πρέπει να δώσουν το καλό παράδειγμα. Σα ευχαριστώ πολύ για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κ. Γκούναρ Χέρτμαρκ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ε, ακούγοντας εδώ τη συζήτηση διαπιστώνει κανείς ένα πράγμα. Νομίζω ότι επικρατεί ευρεία συνένεση επί του ότι χρειαζόμαστε σταθερότητα για να υπάρξουν επενδύσεις και ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή οικονομία. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν είμαστε όλοι σύμφωνοι για το πώς μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό. Ε, βλέποντας όμως το πώς εξελίσσεται η κατάσταση, αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι οι οικονομίες εκείνες ε, οι οποίες τα τελευταία πέντε χρόνια ας πούμε είχαν πολύ καλές προοπτικές ε, για τα επόμενα χρόνια αυτές ε, είχαν σταθερότητα στα δημόσια οικονομικά. Ενώ οι οικονομίες εκείνες που χτυπήθηκαν, επλήγησαν περισσότερο από την κρίση ήταν εκείνες που είχαν αυτό που σήμερα αποκαλείται ευελιξία, δηλαδή είχαν μεγαλύτερα ελλείμματα. Γιατί όσο μεγαλύτερα ελλείμματα έχει κανείς, ε, τόσο μεγαλύτερο βάρος υφίσταται και μεγαλύτερη ανασφάλεια. Ένα σημαντικό πρόβλημα δεν είναι οι οικονομικές πολιτικές ε, σε μεμονωμένα κράτη-μέλη. Υπάρχει και άλλο ένα πρόβλημα που κατά την άποψή μου είναι σημαντικό για όλες τις ε, οικονομίες, ε, ακόμα και για εκείνες που είναι εκτεθειμένες σε ελλείμματα. Δηλαδή, αν βήμα προς βήμα υποσκάπτουμε την αξιοπιστία του Συμφώνου Σταθερότητας, αυτό σημαίνει ότι υποσκάπτουμε τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολό της. Αυτός είναι ένας από τους λόγους γιατί ε, σήμερα υπάρχει σχετική ψυχραιμία στην ευρωπαϊκή οικονομία παρότι γνωρίζουμε ότι μεταξύ βράζουν αρκετά προβλήματα. Επικρατεί λοιπόν η άποψη ότι το σύμφωνο σταθερότητας ε, θα επιφέρει μεγαλύτερη εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών. Και βλέπουμε ότι αρκετά κρατημέλη ακολουθούν αυτόν τον δρόμο και διαπιστώσαμε ότι όσοι το έκαναν τα πράγματα βελτιώθηκαν. Διαπιστώσαμε επίσης ότι η πραγματική λιτότητα εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη που πριν από τη λιτότητα είχαν ε, σπαταλότητα, συσσαγωγικά. Ε, να το πω έτσι, γιατί και στα αγγλικά υπάρχει μια λέξη που είναι ε, και αυτή η πολύ της μόδας, Σπαταλότητα λοιπόν, η οποία... Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι πρέπει να ε, διαφυλάξουμε τη δημοσιονομική εξυγίανση στα κράτη-μέλη, γιατί αυτό είναι προαπαιτούμενο για ε, μακροχρόνιες επενδύσεις και για νέες ε, θέσεις απασχόλησης. Αυτές είναι οι προτεραιότητες λοιπόν, αλλά οφείλουμε να διαφυλάξουμε και το σύμφωνο της σταθερότητας, γιατί αν καταπέσει η αξιοπιστία του συμφώνου σταθερότητας, τότε θα διαλυθούν και πολλά άλλα πράγματα και πολλά θα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς. Thank you very much. Uh, uh Mr. Paolo Guerrieri from Italian Senate. Ο κύριος Γουδιέρη από, από την Ιταλική Σύγκλητο. Ευχαριστώ πολύ. Από την Ιταλική Γερουσία, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Σύγκλητο. Για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Συμφωνούμε ότι η εστίαση της ε, Κομισιόν για το 2016 στις ε, ειδικές αναχώρασης τάσεις είναι ε, ένα από τα κεντρικά στοιχεία. Λοιπόν, οι τρεις πυλώνες των προτεραιοτήτων είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικές. Υποστήριξη των επενδύσεων, διαφορετικές αλλαγές και διατήρηση υγιών και υγιών δημοσίων οικονομικών. Όσον αφορά τις διαφορετικές αλλαγές ε, τις οποίες ε, υλοποιούν ήδη τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον τομέα αυτό μπορεί να ε, υπάρξει σημαντική βελτίωση όσον αφορά και οι ειδικές χώρες και όσον αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιταλία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία μεγάλης προσαρμογής όσον αφορά τις διαφορετικές αλλαγές. Έχουμε υλοποιήσει σχεδόν εξ ολοκλήρου το μεγαλύτερο μέρος των συστάσεων για το 2016 ε, και ε, προχωρούμε, ε, κάνουμε πρόοδο κατά 25% όσον αφορά τις άλλες συστάσεις. Δηλαδή ως χώρα είμαστε απολύτως πεπισμένοι ότι πρόκειται για πολύ σημαντικές δεσμεύσεις. Οπωσδήποτε όμως ε, κάτι ε, επιπλέον θα πρέπει να γίνει από τις μεμονωμένες χώρες, οι μεμονωμένες και της Ιταλίας, όσον αφορά το περιεχόμενο της ε, μεταρρύθμισης. Πρέπει να υπογραμμίσω πάντως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι διευθυντικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε ένα καλό μακροοικονομικό περιβάλλον έτσι ώστε να μπορέσουν ε, να ε, υλοποιηθούν με τρόπο σωστό και αποτελεσματικό. The present economic recovery ε, η οικονομική ανάκαμψη και της ε, ε, ζώνης του ευρώ αλλά και της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ακόμα είναι πολύ χαμηλή. Μετά από πολυετή κρίση και αδυναμία αντιμετώπισης της πολυετούς και ανεργίας. Επομένως καταλαβαίνετε ότι το γενικότερο πλαίσιο δεν είναι ικανοποιητικό. Συμφωνώ βεβαίως με την έκθεση και με τα όσα αναφέρει. Αυτό που είναι ζωτική σημασία τώρα είναι η ανάπτυξη της εσωτερικής ζήτησης στην Ευρωζώνη. Δηλαδή με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να στηρίξουμε την εσωτερική ζήτηση. Είμαστε η πιο πλούσια αγορά ε, στον κόσμο και δεν ε, ε, εκμεταλλευόμαστε αυτή την πλούσια αγορά έτσι ώστε να υποστηρίξουμε την οικονομική ανάπτυξη. Και γιατί αυτό, γιατί ξέρουμε ότι η δημοσιονομική πολιτική δεν υποστηρίζει κατάλληλα την εσωτερική εσωτερική ζήτηση και ακόμα και σε περίπτωση που αυτό γίνεται ε, τα δημόσια οικονομικά δεν, και οι δημόσιες επενδύσεις ε, δεν συμβάλλουν αρκετά. Επομένως, ε, αυτά πρέπει να λάβουμε, η χώρα, να λάβουμε υπόψη μας, έτσι ώστε η χώρα μας να ανακάμψει σε ένα καλύτερο και πιο θετικό περιβάλλον. Επομένως, θα πρέπει να υλοποιηθεί καλύτερη και περισσότερη δημοσιονομική πολιτική. Τι σημαίνει αυτό θα πρέπει να εφαρμόσουμε στην, ε, στο σύνολο της Ευρωζώνης ε, ε, κοινή πολιτική, δημοσιονομική, έτσι ώστε ε, να μπορέσουμε να έχουμε κοινά fiscal stands σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Από το 2011 μέχρι το 2013 αυτή, ε, η, ε, αυτός ο ισολογισμός ήταν αρνητικός. Τώρα, τώρα φτάνει πλέον να γίνεται θετική αυτή η ισορροπία, αλλά δεν συμβάλλει παρόλα αυτά ικανοποιητικά στην ανάκαμψη της οικονομίας. Θα πρέπει να δούμε επομένω τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτήν την ε, νέα δημοσιονομική ε, ε, ισορροπία. Πέρα όμως από τις δημοσιονομικές πολιτικές ε, θα πρέπει να α, μεγαλώσουν, να, να, να αυξηθούν ε, οι δημόσιες ε, επενδύσεις γιατί αυτές μπορούν να συμβάλλουν στη, στη βελτίωση του μικρο και μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Αυτά όσον αφορά το 2017. Thank very much. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ιστβαν από την Ουγγαρία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Εκ μέρου ε, του Ουγγρικού Κοινοβουλίου ε, θέλω να σας ε, ευχαριστήσω και να σας πω ότι τα εθνικά μας κοινοβούλια Ε, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε... Είναι λοιπόν σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι θεωρούμε πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτές οι συστάσεις ανά χώρα, οι οποίες είναι πιο σύντομες, ε, είναι στοχευμένες και αυτό είναι κάτι το πολύ θετικό. Όλα βασίζονται σε ε, πολύ συγκεκριμένες βάσεις και απόψεις και αυτό το βρίσκουμε σημαντικό. Κατά την άποψή μας ε, η σταθερότητα της οικονομίας μας είναι δεδομένη. Σε εμά η οικονομική ανάπτυξη ε, είναι πάνω από το μέσο όρο. Ε, ο προϋπολογισμός στην Ουγγαρία είναι σταθερός και συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ότι η σταθερότητα είναι καθοριστική σημασία για μια χώρα, κυρίως όσον αφορά τα δημοσιονομικά μιας χώρας. Αυτό το κατάλαβε και το αναγνώρισε η Ουγγρική κυβέρνηση. Εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε έλλειμμα κάτω από το 3% και μάλιστα φτάσαμε μέχρι και κάτω από το 2% και όχι μία αρκετές φορές. Γι' αυτό λέμε ότι ο προπολογισμό μας είναι σταθερός. Και εδώ και έξι χρόνια μειώνεται και το χρέος. Και έτσι λοιπόν ε, τα οικονομικά μας είναι υπό έλεγχο. Standard Poor's το αναγνώρισε αυτό και την αξιολόγησε ανάλογα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχοντας επίσης κατά νου και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του 2016, γιατί τα ίδια αποστελέσματα μας τα αναγνώρισε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρούμε ότι ο κίνδυνος ε, ε, ανισορροπίες δεν υπάρχει σε μας ε, στα δικά μας τα δημόσια οικονομικά. Στις συστάσεις αναχώρα της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνονται πολύ συγκεκριμένες προτάσεις με πολύ συγκεκριμένους αριθμούς. Αυτή λοιπόν η παράμετρος για μας πρέπει να παραμείνει και στο μέλλον γιατί μόνο έτσι θα είναι δυνατόν για τα κράτη-μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ε, μόνο δηλαδή εφόσον ε, η Κομισιόν υποβάλλει συγκεκριμένες τεχνικές προτάσεις. Εμείς φέτος έχουμε τρεις ανασυστάσεις χώρα και όχι πέντε που είχαμε στο παρελθόν. Και οι τρεις είναι αποδεκτές για την κυβέρνησή μας. Δημοσιονομική πειθαρχία. Πράγματι θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Κατόπιν, οι ε, φόροι ανατομέα και ανακλάδο. Ε, αυτό προχωράει για να αισθάνονται ε, ασφαλείς ε, οι επιχειρηματίες και περιμένουμε ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις στη χώρα μας. Τα επόμενα χρόνια το πρόγραμμα της οργανωμένης εργασίας θα διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι ε, ενεργοί πολίτες να μπορούν να επανέλθουν το συντομότερο δυνατόν στην αγορά εργασίας. Εν ολίγης, εμείς ε, σεβόμεθα και δεχόμεθα τις ανασυστάσεις χώρα Πριν από δύο περίπου χρόνια είχαμε στην Ουγγαρία τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τον, είχαμε και το Γενικό Διευθυντή ε, Υποθέσεων, μιλήσαμε για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα και μιλήσαμε και για τις ανασυστάσεις χώρα. Σε γενικές γραμμές λοιπόν τις ε, αλλαγές... Ε, τις ε, θεωρούμε θετικές και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υλοποιηθούν οι αλλαγές αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Μπαλάουρας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκουλτιέρη, χαίρομαι που σας γνωρίζω και προσωπικά. έχουμε ανταλλάξει ορισμένα μηνύματα σας θεωρώ έναν άνθρωπο ε, αντικειμενικό, έναν άνθρωπο που δεν διστάζει να πει την άποψή του ε, που τελικά καταγράφεται σαν ένας φίλος της χώρας μας, της Ελλάδας και νομίζω ότι έχουν την άποψη αυτή και όλοι, όχι μόνο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ε, η χώρα μας, όπως ξέρετε, είναι ε, σε ένα ε, πλαίσιο ε, στήριξης που άμεσα δεν συμμετέχει στην, στο πρόγραμμα που συζητιέται σήμερα εδώ. Όμως αυτή η πολιτική που σήμερα συζητάμε αντικειμενικά επηρεάζει όχι μόνο τα κράτη που δεν είναι ε, σε πρόγραμμα, αλλά και τα κράτη που είναι στο πρόγραμμα όπως η χώρα μας. Επομένως, πρέπει να δούμε τα αίτια της οικονομικής κρίσης εν συνόλο. Γιατί άραγε όταν μαζί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι, και οι Ηνωμένε Πολιτείε μπήκαν σε κρίση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε εδώ και τρία περίπου χρόνια έχουν βγει και μάλιστα με ψηλού ρυθμούς ανάπτυξης τι άραγε φταίει στην ασκούμενη οικονομική πολιτική. Άκουσα συναδέρφους ήδη που μίλησαν που αναφέρθηκαν στις μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις προς τι και σε ποια κατεύθυνση. Δεν είναι ουδέτερες έννοιες αυτές. Είναι γνωστό ότι η Ευρώπη κυριαρχείται από τον νεοφιλελευθερισμό. Επομένως, μεταρρυθμίσεις με διάλυση του κοινωνικού κράτους μεταρρυθμίσεις με απελευθέρωση της αγοράς εργασίας χωρίς δικαιώματα στους εργαζόμενους. Να τα δούμε λοιπόν αυτά. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση λέγοντας με όρους γνωστούς από την οικονομία ορισμένα πράγματα. Η εκτίμηση, συνάδελφοι, των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε φεσιακό κράχ. Όπως θα έλεγα όχι του 29 στις, που αγκάλιασε όλη την, ε, το, όλη την, ε, ε, τον κόσμο, αλλά το τελευταία χρόνια την Ελλάδα. Η εκτίμηση λοιπόν, το ξαναλέω, των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε φυσιακό κράχ. Η ανάπτυξη, και εδώ είναι μια περίεργη λέξη που θα πω, είναι σε ύφεση. δεν υπάρχει ανάπτυξη, το αντίθετο υπάρχει πανάπτυξη. Η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε σασιμότητα. Αύξηση με υψηλό μάλιστα πολλαπλασιαστή στις ανισότητες, δηλαδή στο κοινωνικό περιβάλλον συνολικά αλλά και στο περιφερειακό. Και ταυτόχρονα έχουμε boom στη φτώχεια και στην ανεργία. Για παράδειγμα, δεν θέλω να αναφέρω την Ελλάδα τόσο, αλλά απλώς να σας το ξαναθυμίσω, τα τελευταία χρόνια αυτής της ε, θεραπείας για την Ελλάδα. Η, η ανεργία έχει φτάσει στο 27% έτσι. και πολλά άλλα πράγματα. Το κρέος έχει υπερδιπλασιαστεί ε, και δεν έχουμε βγει ακόμα από την κρίση. Επομένως, συνάδελφοι, νομίζω ότι χρειάζεται μια αλλα... ριζική αλλαγή αυτή του ε, πλαισίου. Να υπάρξει ένα σύμφωνο ανάπτυξης ένα σύμφωνο το οποίο θα μιλάει για βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη με δικαίωμα στην εργασία και στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που σήμερα παραβιάζονται. Πρέπει ταυτόχρονα να ενδυναμωθεί ο διάλογος με τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωκοινοβούλιο και να υπάρξει μια ουσιαστική ενίσχυση των κοινωνικών δικτών. Θα το έλεγα και με άλλη φρασολογία ότι η ανεργία και η φτώχεια στις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ανεξάρτητες μεταβλητές που χρειάζονται αντιμετώπιση με συγκεκριμένε πολιτικές αλλά παρεπόμενες άλλων πολιτικών που θεωρούνται κεντρικές όπως για παράδειγμα η δημοσιονομική σταθερότητα. Ο πολίτης, ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος χάνεται σε τέτοιες εκφράσεις οι οποίες κατά τη γνώμη μου βαλτώνουν ακόμα περαιτέρω την ευρωπαϊκή οικονομία και τα επιμέρους κράτη και ε, χάνει τη φερεγγιότητά της, ήδη την έχει χάσει αρκετά, χάνει αυτή τη λάμψη που είχε από την είδηση της Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ξέρω πού θα οδηγήσει μετά και από τον Brexit που πρόσφατα ζήσαμε και ζούμε τα αποτελέσματά τους και μάλιστα είναι η αρχή των αποτελεσμάτων. Και, μάλι, και εδώ θέλω να τονίσω επίσης ότι υπάρχουν και δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η, η Γερμανία για παράδειγμα έχει ένα πλεόνασμα του 8% το οποίο δεν είναι συμβατό με τις ε, ευρωπαϊκές συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ ε, που με ακούσατε και νομίζω ότι θα γίνει ένας ενδιαφέρον διάλογος ε, για αυτά τα ζητήματα. Thank you. Mr. Σας ευχαριστώ πολύ. 9%. Είπατε 9%. Yes, it's, it's more. Ναι, 9%. Πρωτογενές. Η κυρία Περβόνς Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, είναι πάρα πολύ καλό που έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων, γιατί είναι η στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να συζητήσει τις ειδικέ συστάσει, αλλά και γενικότερα την αναπτυξιακή πολιτική ε, για το επόμενο έτος. Και επομένω είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων, γιατί ε, ο τρόπος υλοποίηση επίσης των ειδικών αναχώρα συστάσεων είναι μια εξαιρετικά επίπονη και συγκεκριμένη εργασία. Ε, ακούμε και δηλώσεις, ακούμε και διεκδικήσεις από την πλευρά των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, και ε, για να είναι οι συστάσεις ε, ολιγαριθμές αλλά καλύτερα συντονισμένες με την πραγματικότητα της κάθε χώρας και όχι να υπάρχει απλώς ένα copy-paste για όλες τις χώρες. Αυτό υπόθηκε και υπογραμμίστηκε. Ε, κοιτάξτε, οι ειδικέ συστάσεις αναχώρα σημαίνουν ε, και κάποιες ε, ε, οικονομικές ας πούμε συστάσεις ή αναφέρονται, πώς να σας το πω ευγενικά, αναφέρονται σε κάποιες οικονομικές πολιτικές οι οποίες για να προοδεύσουν χρειάζεται ακόμα μεγάλη προσπάθεια, να το πω έτσι πιο ευγενικά. Η χρήση του συνόλου των εργαλείων ε, που έχουμε ε, στη διάθεσή μας ε, όσον αφορά την οικονομική πολιτική, η χρήση λέω όλων αυτών των εργαλείων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, αυτή η Microeconomic Imbalance Procedure, η MIP, ε, χρησιμοποιείται. Αλλά βέβαια πρέπει να δούμε όλες, ε, όλα τα συμπεράσματα τα οποία μπορούν να απορρεύσουν από αυτήν την παρατήρηση της MIP. Είναι λύση για όλα. Δεν το πιστεύω εγώ προσωπικά. Και νομίζω ότι όταν η Κομισιόν βάσει του 2 pac και του 6-pack ζητά να γίνουν σεβαστοί οι κανόνες, κανόνες ε, θα πρέπει, ε, και είναι πολύ αυστηρή, θα πρέπει η Κομισιόν να σκεφτεί ότι την ίδια αυστηρότητα θα πρέπει να ζητήσει για την εφαρμογή και όλων των άλλων κανόνων. Και νομίζω ότι και εδώ μπορεί να έχουμε κάποιο περιθώριο βελτίωσης. Δεύτερον, το θέμα των επενδύσεων. Η Κομισιόν ορθώς ε, ε αναφέρεται εδώ εξειδικευμένα αλλά κάποιος ομιλητής, δεν θυμάμαι ποιο, αναφέρθηκε ε, στη διαφοροποίηση ανάμεσα σε επενδύσεις ε, δημόσιες ε, και ιδιωτικές. Ξέρουμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, η εμπιστοσύνη δεν έχει αποκατασταθεί πλήρω, άρα θα πρέπει λίγο να βασιστούμε και στα δύο αυτά σκέλη, και στι δημόσιε και στι ιδιωτικές επενδύσεις. Μη λησμονούμε ότι βρισκόμαστε στη στιγμή κατά την οποία συζητούμε τη δεύτερη φάση ε, τη, του, του προγράμματος Juncker και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να ε, δημιουργήσουμε αυτό το ε, πρωτόλιο ας πούμε ε, εργαλείο μακροοικονομικής πολιτικής και να δούμε και να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε και πώς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το νέο σχέδιο Juncker έτσι ώστε να μπορέσουμε να σηκώσουμε τον πύχη στις οικονομίες μας. Τρίτον, Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος ε, να αναφερθούμε, ε, να πάμε πολύ μακριά όταν ε, αναφερόμαστε στις ειδικέ συστάσεις αναχώρα. Δηλαδή, πιστεύω ότι υπάρχει ένας χώρος που μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο όσον αφορά τα δημοσιονομικά. Στον τομέα των δημοσιονομικών ξέρουμε ότι δεν είναι πλήρης αρμοδιότητα σε ενωσιακό επίπεδο, αλλά ακριβώς μέσω αυτών, αυτές οι αναχώρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια καλή ευκαιρία ε, συνολικής διαιτησίας κατά κάποιο τρόπο όσον αφορά αυτά, αυτές τις δημοσιονομικές πολιτικές. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει ε, στις συστάσεις αυτές μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στη δημοσιονομική αντιμετώπιση του κεφαλαίου και της εργασίας. Και αυτός θα πρέπει να είναι ένας κοινός στόχος. Thank you, Ευχαριστώ πολύ. Πάολο Τίνκο Περέιρα από την Πορτογαλία. Grazie, signor Presidente. Members of European Parliament. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων. Θέλω να σας πω ότι είμαι το μόνο μέλος του Πορτογαλικού Κοινοβουλίου που βρίσκομαι εδώ σήμερα και θα προσπαθήσω να σας ε, μεταφέρω ε, αυτό που επί συμφωνούν όλοι οι κοινοβουλευτικοί στην Πορτογαλία και συμφωνούν γενικότερα περισσότεροι στη χώρα μου. Αυτή η συνάντηση έρχεται σε μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή. Όπως ε, ξέρετε, στις 3 Οκτωβρίου θα υπάρξει μια ε, κοινή συνάντηση της ΕΚΟΝ και της ε, ΡΕΤΖΙ και των Επιτρόπων Καϊτάνεν και Κρετή. Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται ο περίφημος διαρθρωμένος διάλογος ανάμεσα στην Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα αυτής της συνάντησης, όπως γνωρίζετε ορισμένοι ημών, είναι ότι ε, θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις ε, στην Ισπανία και την Πορτογαλία, να τους ανασταλούν ε, οι κάποια κονδύλια, γιατί οι δύο αυτές χώρες το 2015 δεν εφάρμοσαν πλήρως τις συστάσεις της Κομισιόν. Δύο μηνύματα λοιπόν θέλω να εκφράσω σήμερα. Το ένα είναι ότι υπάρχει ομόφωνη συνένεση όσον αφορά ένα ευρύ πολιτικό φάσμα. Και θέλω να πω όσον αφορά και την πλειοψηφία των Πορτογάλων πολιτών ότι αυτές οι κυρώσεις όχι μόνο είναι άδικες αλλά είναι και αντιπαραγωγικές. Η απόφαση επιβολής κυρώσεων ε, θα μειώσει την ε, υποστήριξη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στην Πορτογαλία. Γνωρίζω ότι σε όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς υπάρχουν οι περίφημοι σκληροπυρηνικοί που λένε ότι οι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τις οικονομικές συνέπειες. Και υπάρχουν και οι άλλοι που θεωρούν ότι οι κανόνες είναι το μέσο για να επιτύχει κανείς το στόχο του, άρα θα πρέπει να ερμηνεύονται με κάποια ευελιξία, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες όχι μόνο σε μια συγκεκριμένη χώρα, αλλά και όσον αφορά στην αξιοπιστία των των ίδιων των κανόνων. Ως εκ τούτου, το δεύτερο μήνυμα που θέλω να σας εκφράσω είναι ότι εμείς ε, εφαρμόζουμε τους ε, κανόνες με κάποια ευελιξία. Ο δικός μου στόχος είναι η σκληροπυρηνική. Να τους πείσω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που συμφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Ε, ποιο είναι στο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα το σημαντικό είναι ε, να παραμείνουν μετά το Brexit όλα τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από ένα χρόνο αυτό δεν ήταν στόχος και είχαμε υποθέσει ότι ε, Σήμερα αυτός είναι ένας στόχος που πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένας βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να σας πω ε, τι ακριβώς αναφέρεται στην ετήσια έρευνα. Ένα από τα βασικά θέματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος είναι να προάγει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος ε, ε, προτεραιότητας, η πρώτη προτεραιότητα ε, εδώ πρέπει να αναφέρω ότι η Τραπεζική Ένωση πρέπει να ολοκληρωθεί για να υπάρχει μεγαλύτερη δημοσιονομική σταθερότητα. Χωρίς λοιπόν ανάπτυξη και απασχόληση, το ευρωπαϊκό εγχείρημα θα αποτύχει. Ε, δεν έχω χρόνο για να μπω σε λεπτομέρειες. Ίσως θα ολοκληρώσω και ελπίζω να μου δοθεί κάποιος έξτρα χρόνος αργότερα. Να σας πω με λίγα λόγια ποια είναι η κατάσταση στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία θα ξεφύγει από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος το 2016. Αυτή είναι η πρόβλεψη της Κομισιόν. Τώρα έχουμε έλλειμμα 2,7%. Άρα εμείς ε, εφαρμόζουμε ε, δημοσιονομική εξυγίανση. Και το θέμα που τίθεται επιτάπτως είναι κατά πόσον θα πρέπει να τιμωρηθεί μια χώρα η οποία προβαίνει σε δημοσιονομική εξυγίανση, σε ανάπτυξη και απασχόληση. Και ελπίζω ε, να μπορέσω σε λίγο να επανέλθω για να σχολιάσω αυτά τα θέματα. Ευχαριστούμε πολύ. Next uh, Ευχαριστώ που μας υπενθυμίσατε ότι την άλλη Δευτέρα θα έχουμε αυτόν τον δομημένο διάλογο στην Επιτροπή Οικονομικών και Περιφερειακής Πολιτικής με τους Επιτρόπους Κατάνιν και Κρέτσου για την ε, πιθανότητα αναστολής των διαρθρωτικών τομείων. Θα είναι σημαντική η συνεδρίαση και σημαντική και η παρέμβασή σας. Η θέση της Πορτογαλίας για το θέμα αυτό. Μάρκο Βάλλη, το EFTD. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι ήρθαν εδώ για τον διάλογο. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι αυτό το ευρωπαϊκό όνειρο τελικά έχει μετατραπεί σε φιάλτη. Γιατί υπάρχουν αυτές οι συστάσεις ε, που δίδονται στις ε, χώρες που δεν αρέσουν όμως ε, ούτε στους πολίτες ούτε στους εκπροσώπους των πολιτών. Γιατί είναι μια συνταγή η οποία έχει αποτύχει. Δηλαδή λιτότητα, ιδιωτικοποίηση, ιδιωτικές επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις, μειώσεις μισθών μέσω των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασία, αυτά στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Πορτογαλία και γιατί εφαρμόζονται όλα αυτά για να υπερασπιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση το ευρώ γιατί ε, αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν νομισματικές διακυμάνσεις επειδή υπάρχει σταθερό νόμισμα αλλά το μόνο που υπάρχει είναι να ε, περικόπτονται μισθοί. Αυτό αναφέρθηκε και αυτό το καλοκαίρι, ότι δεν βάζουμε το δάχτυλο στο πρόβλημα το πολιτικό που είναι η νομισματική ένωση, αλλά ε, βλέπουμε ότι η, τελικά η νομισματική ένωση αφορά 19 χώρες. Όμως οι 19 χώρες δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες. Έχουν διαφορετικές ανάγκες παραδείγματο χάρη των επιτοκίων. Και δεν αντιμετωπίζουμε το γεγονός ότι έχουμε 24 διαφορετικές γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό και μόνο το γεγονός περιορίζει την κινητικότητα των εργαζομένων. Στι ΗΠΑ υπάρχει μία μόνο γλώσσα και εκεί υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες για τους εργαζόμενους να μετακινηθούν. Ε, αυτό δεν ισχύει λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου υπάρχει κάποια αντίφαση. Το είπα αυτό και στον Τράγκη και σε άλλους οικονομολόγους οι οποίοι δεν εγκρίνουν αυτό που κατά την άποψή μου είναι ένα πρόγραμμα που δεν οδηγεί πουθενά. Είτε θα αλλάξουμε ε, το, το πρότυπο που εφαρμόζουμε, που θεωρούμε το ευρώ ε, ιερό και όσιο ή σε τελική ανάλυση θα έχουμε ακόμα χειρότερη κατάσταση γιατί θα φτάσει κάποια στιγμή όπου ε, κάποια κράτη θα τελείσουν μονόπλευρα και με δική τους ευθύνη να φύγουν από το ευρώ. Αυτά που αναφέρθηκαν και που επιβάλλονται εξάλλου δεν είναι δημοκρατικά. Είδαμε τι γίνεται στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Οι δύο χώρες δεν συμφωνούν. Ε, δεν συμφωνούν το να δεχθούν ε, τιμωρία και κυρώσει. Ε, δεν μπορούν οι πολιτικοί που εκπροσωπούν αυτές τις χώρες ε, να κάνουν οτιδήποτε αν δεν συμφωνήσουν οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το πρόγραμμα κατά την απόψή μου δεν μπορεί κανείς να το υπερασπιστεί και είναι και πολύ επικίνδυνο ε, γιατί τελικά γυρίζουμε γύρω γύρω από το πρόβλημα. Τα προβλήματα που αφορούν στην αναθεώρηση της διακυβέρνησης αυτά δεν είναι και πολύ σοβαρά γιατί έχουμε ας πούμε τον, ε, την πρόταση για έναν Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομικών ή θεσμοθέτηση της Τρόικα, δηλαδή να είναι ένας εμπειρογνώμονας ο οποίος θα παίρνει τα χρήματά σας από τον προπολογισμό και θα σας λέει πώς να εφαρμόζετε τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό ε, θα πρέπει να το εξηγήσετε στους ε, ψηφοφόρους αν υιοθετήσετε αυτή τη γραμμή. Είναι πολύ δύσκολο να υιοθετήσει κανείς αυτή τη γραμμή. Είναι πολύ πιο εύκολο να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα και να συνεχίσουμε τη συνεργασία μα γιατί αλλιώς θα καταλήξουμε στο να έχουμε μία ανεξέλεγκτη διάλυση, κερδοσκοπία, θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα επενδύουν στην ευρωπαϊκή σύγκρουση και νομίζω οι περισσότεροι αντιευρωπαίοι αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς αυτοί οι εμπειρογνώμονες οι οποίοι ε, προσπαθούν να εφαρμόσουν ε, αρχές οι οποίες όμως αποδείχθηκε ότι έχουν αποτύχει τα τελευταία χρόνια και υπάρχει σε να ζήσουμε μια κρίση χωρίς προηγούμενο αν δεν σταματήσουμε να υπερασπιζόμεθα ε, χωρίς φραγμούς αυτό το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία Ήτανε πολλές φορές στην υπηρεσία πολλών άλλων δυνάμεων. Οι πολίτες μας ρωτάνε, μα τι κάνετε, ποιους εκπροσωπείτε. Ε, αυτή είναι η ευχή μου. Εγώ εκπροσωπώ μια νέα πολιτική δύναμη στην Ιταλία. Ε, στις σφιγμομετρήσεις όμως είμαστε πρώτοι. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι προσπαθούμε και εμείς να σας ταρακουνήσουμε για να περάσουμε σε μια νέα μορφή ε, συνεργασίας γιατί αλλιώς ε, συνεργαζόμαστε με άτομα που θα μας οδηγήσουν στην καταστροφή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ονόφριος Κούλας από την Κύπρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, αισθανόμαστε ευτυχεί που επανεντασσόμαστε στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος προσαρμογής που εφαρμόσαμε και που ε, ολοκληρώσαμε τον περασμένο Μάρτιο. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θεωρούμε ότι είναι μια σημαντική διαδικασία καθότι καθορίζει το πλαίσιο διαλόγου για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο και θα τονίσω το σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί και εκεί χρειαζόμαστε πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Ε, είναι γνωστό ότι η ζώνη του ευρώ είναι μια ατελής νομισματική ένωση και χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να αφαιρέσουμε όσο γίνεται αυτή της ατέλης. Επίσης, με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο εντοπίζονται οι μακροοικονομικές ανισορροπίες σε κάθε κράτος μέλος, ε, οι οποίες είναι όντως δυνατόν να εξαχθούν σε άλλα κράτη-μέλη και οι συστάσεις που γίνονται για κάθε χώρα είναι πιστεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο συντονισμός των πολιτικών μας, μια πιο ενοποιημένη Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγματι πιστεύουμε ότι θα προσθέσει αξία στην επίτευξη των κοινών μας στόχων. Όσον αφορά τις ειδικέ συστάσεις για την Κύπρο, θα πρέπει να πούμε ότι συμφωνούμε με αυτές. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στα πλαίσια του προγράμματος προσαρμογής, όπως για παράδειγμα με το συνταξιοδοτικό, αλλά ε, έχουμε επίσης ε, εισαγάγει και ένα ελάχιστο εγκυημένο εισόδημα για κάθε οικογένεια και για κάθε πολίτη που έχει ανάγκη εκείνη την ώρα. Ε, Άρα δεν είναι απλά μεταρρυθμίσεις ε, κατά ανάγκη βάρος των εργαζομένων ή των πολιτών, μπορεί να είναι και μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση που όπως αντιλαμβάνουμε οι περισσότεροι θα ήθελαν. Η κυβέρνηση μας έχει ήδη καταθέσει αρκετά νομοσχέδια τα οποία συζητούμε αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Κοινοβούλιο για να και ελπίζω ότι πολύ σύντομα πριν το τέλος του χρόνου θα ψηφιστούν σε νομοθεσίες. Αυτά αφορούν, για παράδειγμα, την μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, την κινητικότητα των υπαλλήλων, από κάθε τμήμα, από κάθε Υπουργείο και με, με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έτσι ώστε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα. Συζητάμε επίσης για μεταρρύθμιση των τοπικών κυβερνήσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης έτσι ώστε υποχρεωτικά να έχουν ε, κοινέ υπηρεσίε προ όφελο του πολίτη στο χαμηλότερο δυνατό κόστο. Συμφωνούμε επίση και αναγνωρίζουμε τις ε, μακροοικονομικέ ανισορροπίε που έχουν εντοπιστεί, όπω το υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέο, καθώς και το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο τραπεζικό σύστημα. Πέραν των ειδικών ενεργειών που γίνονται για να αντιμετωπιστούν ε, όλοι αυτοί οι κίνδυνοι, θα πρέπει να πω ότι η καλύτερη από το αναμενόμενο απόδοση της οικονομίας μας κάνει πολύ αισιόδοξου. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις, για το 2016 αναμένουμε ρυθμό ανάπτυξης που θα ξεπεράσει το 2,7%. Είναι πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έχουμε περίπου μηδενικό δημοσιονομικό έλλειμμα. Ε, θα είναι σχεδόν 0%. Τα ίδια αποτελέσματα και καλύτερα περιμένουμε με τον προπολογισμό του 2017 ότι η ανάπτυξη θα ξεπεράσει ή θα είναι πολύ κοντά στο 3% και το δημοσιονομικό έλλειμμα θα είναι το πολύ μισό της εκατό του ΑΕΠ. Ε, με αυτά πιστεύουμε ότι το δημόσιο χρέος, το ιδιωτικό χρέος, η ανεργία και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που βαίνουν ε, μειούμενα θα, θα επιταχυνθεί αυτή η μείωση. Ε, αυτό το μικρό δημοσιονομικό περιθώριο που είχαμε μας έδωσε και την ευχαίρεια να μειώσουμε στοχευμένα κάποια τέλη ή φορολογίες που θα εθαρρύνουν τις επενδύσεις από τούτα και στο εξή. Ξέρετε, θα κλείσω με το εξή. Θα πω ότι ε, είναι ένα καλό παράδειγμα αυτά τα αποτελέσματα πώς μπορείς να έχεις δημοσιονομική ισορροπία και ανάπτυξη ταυτόχρονα. Πήραμε σκληρά μέτρα όντω και δημιουργήσαμε ύφεση για μια διετία. Εξαλείψαμε όμω το δημοσιονομικό έλλειμμα από 6% σε 0% σε μία διετία και από τούδε και στο εξή προχωράμε με ένα βιώσιμο ρυθμό ανάπτυξη, τον οποίο πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε σύμφωνα με τι προβλέψει μέχρι και το 2020 τουλάχιστον. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ρίχαρτς Κόλτς από την ε, Λετωνία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω, δεν θέλω να προσθέσω τίποτα για το CSR, αλλά θέλω να εστιάσω την προσοχή μου σε ένα συγκεκριμένο θέμα που κατά την άποψή μου ε, δεν έχει εξεταστεί μέχρι σήμερα και είναι ένας από τους λόγους ε, γιατί έχουμε τόσο χαμηλή οικονομική ανάπτυξη. Και μάλιστα αυτό επηρεάζει και το καθήκον μας που είναι να αντιμετωπίσουμε την γκρίζα οικονομία. Αναφέρομαι στην λατρέα απασχόληση που μπορεί να είναι μέχρι το 7% του ΑΕΠ και προκαλεί ε, πολλές ε, παρενέργειες. Επηρεάζει το σύστημα της ε, κοινωνικής ευημερίας, τα δημόσια οικονομικά. Γιατί λοιπόν αυτό το συγκεκριμένο θέμα δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο της έκθεσης. Κοιτάξτε, η νόμιμη απασχόληση έχει κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Αυτό συνδυάζεται με την μετανάστευση που έχουμε τώρα στην Ευρώπη. Έχουμε στοιχεία από τη Γερμανία ότι 500 ετούντες άσυλο ε, μένουν εκεί παρότι δεν τους προσφέρεται ε, προστασία. Άρα από τι ζουν αυτοί και αυτό απαιτεί από τους ε, πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρουν κάποια θέση απασχόλησης. Ίσως λοιπόν υπάρχουν και κάποια κίνητρα να αντιμετωπιστεί η παράτυπη απασχόληση στα κράτη-μέλη. Αυτό απασχολεί και τη Λετωνία και είμαι σίγουρος ότι απασχολεί και άλλα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ταρπάτη. Äh, ναι. Εγώ είμαι για το ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Ακούστηκαν ήδη κάποια σημαντικά, σημαντικές κουβέντες, ανάπτυξη, επενδύσεις. Ο Έλληνας συνάδελφος είπε πως χωρίς οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτύχει. Πράγματι σκληρό, αλλά είναι η αλήθεια. Πρέπει να δούμε τα πράγματα λοιπόν, πώς έχουν. Υπάρχουν ε, λόγοι και είναι περισσότερο η Ευρωζώνη παρά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωζώνη λοιπόν δεν είναι ενιαία αλλά είναι διχασμένη. Έχουμε παραδείγματο χάρη ε, άνηση εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας. Αν δούμε παραδείγματο χάρη την Ευρωζώνη ως κομμάτι της παγκόσμιας, της, της παγκόσμιας οικονομίας η Κίνα αυξήθηκε, το μερίδιο της Γερμανίας έμεινε σταθερό, η Γαλλία και η Ιταλία μειώθηκαν ως ποσοστό στο μισό σχεδόν του παγκοσμίου ΑΕΠ, οπότε μειώνονται οι εξαγωγές και άρα δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Αν δούμε λοιπόν την ε, ανάπτυξή μας, το προβλέπεται για την Ευρωζώνη 1,6%. Η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με συγχωρείτε, χωρίς Ευρωζώνη, είναι 2,7%. Και αν ε, ε, βγάλουμε τις ε, κάποιες χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ακόμη πιο καταθλιπτικά τα νούμερα. Πρέπει να ρωτήσουμε γιατί είναι έτσι τα πράγματα, γιατί η Ευρωζώνη είναι το κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας που αναπτύσσεται λιγότερο. Αυτό είναι. Ποια είναι η αιτία λοιπόν. Σε τι οφείλεται το ότι στην ε, Γερμανία από το 2010 η ανεργία πήγε από το 10% στο 5% που οφείλεται στο το ότι η ανάπτυξη σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης, στο Νότο, είναι διαφορετική. Η ανεργία από το 10% πήγε στο 25% στο 30% τεράστια. Ποια είναι η αιτία Κοιτάξτε, κάποιοι θα έλεγαν ότι είναι λανθασμένη ισοτιμία. Αν το νόμισμα αυτό είναι υπερτιμημένο για τις χώρες του Νότου και υποτιμημένο για τη Γερμανία και τις άλλες χώρες, ε, είναι σαφές ότι θα έχουμε τέτοιες εξελίξεις. Επιδοτούνται οι εξαγωγές από τη Γερμανία. Δεν χρειάζεται λοιπόν να κοπιάσουν πολύ για να εξάγουν. Ε, αντιθέτως φορολογούνται οι εξαγωγέ από τις χώρες του Νότου. Όταν είναι δηλαδή το νόμισμα υπερτιμημένο, ε, τότε έχουν δυσκολίες. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Ε, και προσπαθεί ο κύριος Ντράγκη με μηδενικά επιτόκια, με αρνητικά επιτόκια. Δεν γίνεται τίποτα. Καμία νομισματική πολιτική δεν μπορεί να ε, εξαλείψει τελείως το πρόβλημα αυτό. Και δεν μπορεί ε, επίσης να κάνει κάτι για το ότι οι δύο αυτοί πόλοι αποκλίνουν. Δεν, ανάγκη να, δεν αρκεί να λέμε συνεχώς χρειαζόμαστε ανάπτυξη. Γιατί έχουν άλλες χώρες μεγαλύτερη ανάπτυξη από εμάς εδώ. Αν απαντήσουμε αυτή την ερώτηση τότε θα καταλήξουμε σωστό συμπέρασμα. Αλλιώ και του χρόνου και του παραχρόνου, κύριε Πρόεδρε, θα έχουμε συνεχώς τα ίδια προβλήματα. Ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερες επενδύσεις, δημόσιες, ιδιωτικές. Μα ο κάθε επενδυτής κοιτάει σε κάθε χώρα ποιε είναι οι προοπτικές, οι μελλοντικέ. Αν οι προοπτικέ δεν είναι καλέ, εμεί μπορεί να λέμε ότι θέμε εδώ μέσα για την αναγκαιότητα δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων. Δεν θα γίνει τίποτα. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κλάουδιο από τη Μάλτα. Χωρίς μικρόφωνο, παρακαλούμε το μικρόφωνο σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ τον συνάδελφο ε, Σάντα για την ε, έκθεση την οποία έκανε και όπου αναφέρει όλους αυτούς τους τομείς που και συνδέονται μεταξύ τους και είναι απαραίτητοι έτσι ώστε να υπάρξει ανάπτυξη στην Ευρώπη. Αναμφίβολα οι τρεις ε, κύριες ε, πρωτοβουλίες ε, της, της Κομισιόν για την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής οικονομίας αποτελούν σωστή βάση και αυτό αποδεικνύεται και από τη συζήτηση. Εγώ θα ήθελα να εστιαστώ περισσότερο στην πρώτη ε, προτεραιότητα, δηλαδή την υποστήριξη των επενδύσεων και πρέπει να πω ότι ε, ε, εάν θέλουμε, αν δεν αλλάξουμε καθόλου την νομισματική πολιτική, οπωσδήποτε δεν θα μπορέσουμε να έχουμε επιτάχυνση των επενδύσεων. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει ε, να δοθεί πολύ μεγαλύτερη προσοχή σε αυτήν την ανάκαμψη, την αναπτυξιακή. Και ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εστιάσουμε την προσοχή μας στην καινοτομία. Η καινοτομία φέρνει προστιθέμενη αξία, η οποία επιταχύνει την παραγωγικότητα και ε, που αυτή μεταφράζεται σε ανάπτυξη και βιώσιμη δραστηριότητα. Διαφορετικά το ε, αποτέλεσμα δεν θα είναι ε, περισσότερες ε, θέσεις. Με τη γενοτομία θα έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και καλύτερες επιδόσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως σε κρίζωση της ένδυας. Κατά αυτή την έννοια θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες έτσι ώστε να αναπτυχθεί η καινοτομία, όχι όμως από πάνω προς τα κάτω, αλλά μάλλον αντίθετα, ανάποδα, από κάτω προς τα πάνω. Επίσης πρέπει να πω ότι θα πρέπει να ε, δώσουμε, ε, να εγχύσουμε κατά κάποιο τρόπο στη ρόλη διαδικασία μεγαλύτερη έννοια ε, αλληλεγγύης, προγράμματα, πλαίσια τα οποία τα οποία θα δημιουργήσουν ένα καλύτερο πλαίσιο για την καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρώπη και διαμέσου της Ευρώπης. Ειδικά δεν αναφέρομαι στις χώρες μέλη, οι οποίες ε, είναι ε, ουραγοί όσον αφορά την καινοτομία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Η Παλώμα Λόπες από την Γκουε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μιλάμε για συστάσεις, ε, ενώ αυτό που πρέπει να λάβει η χώρα είναι ε, ριζική αλλαγή των πολιτικών που εφαρμόζονται. Χρειαζόμαστε ε, διαφορετική φορολογική και βαθμιαία φορολόγηση. Χρειαζόμαστε δημόσιες επενδύσεις. Τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που γίνονται. Θυσιάζουμε τους λαούς μας σε μια νομισματική πολιτική η οποία δεν δίνει αποτελέσματα, δεν λειτουργεί. Αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών, ούτε την ανισότητα, ούτε την ανεργία. Ε, αυτά είναι αποτελέσματα των νέων φιλελεύθερων πολιτικών. Ε, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανάπτυξη μέσα από διασώσεις ε, τραπεζικών συστημάτων. Εμείς δεν είχαμε χρέος, τώρα έχουμε διπλασιασμό του χρέους με ταυτόχρονη κατακρίμνηση του ΑΕΠ. Ε, όλα αυτά τα πλήρωσαν οι εργαζόμενοι. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για διατήρηση των κοινωνικών δικαιωμάτων ενώ δημιουργούμε ένα πλαίσιο το οποίο ευνοεί τις μετακινήσεις ε, των επιχειρήσεων από τη μία χώρα στην άλλη δημιουργώντας μια καταστροφική αλυσίδα. Οι συστάσεις οι οποίες ε, προτείνονται στην ουσία βαθαίνουν ακόμα περισσότερο την κρίση και τις κοινωνικές επιπτώσεις που έχει και εφαρμόζονται με τον εκβιασμό των ε, κυβερνήσεων όσον αφορά την μείωση ή την πάυση της χρηματοδότησης. Επίσης βαθαίνουν οι διαφορές ανάμεσα σε χώρες. Ε, η Γερμανία ή η Ολλανδία μπορεί να έχουν ε, υπερβολικά... Έχουν υπερβολικά πλεονάσματα, ενώ αντίστοιχα οι άλλες χώρες έχουν υπερβολικά δημοσιονομικά ε, ελλείμματα. Ε, ε, στην ουσία αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι μερικέ χώρε απλώ γίνεται προσπάθεια να τι κατακριμνήσουμε, να τι καταποντήσουμε ακόμα περισσότερο. Κρέμεται μία δαμόκλια σπάθη πάνω από χώρε όπω η Πορτογαλία ή όπω η Ελλάδα και μπορώ να δώσω και άλλα παραδείγματα. Πώ είναι δυνατόν να ελπίζουμε ότι οι πολιτικέ τι οποίε αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν καμία σχέση με την εθνική κυριαρχία και τη δημοκρατία. Η, η, η, κυβέρνηση ε, παρουσίασε χωρίς να τους περάσει πρώτα από το κοινοβούλιο της χώρας τις νέες ε, οικονομικές πολιτικές της χώρας και τις υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει έτσι. Πρέπει να χτίσουμε μια άλλη Ευρώπη. Very Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Σίλβα Περέιρα. Obrigado, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω ένα σύντομο σχόλιο για να πω ότι αυτή τη βδομάδα το, στην Επιτροπή ΕΚΟΝ υποδεχτήκαμε τον πρόεδρο της ε, Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος μας, έκανε, μας έδωσε κάποιες ε, προοπτικές ε, για την ανάπτυξη στις χώρες της Ευρωζώνης και ότι μας είπε ότι προσδοκεί ότι η ανάπτυξη θα ξεπεράσει τις πρώτες εκτιμήσεις και θα φτάσει στο 1,6 για το 2018. Επίσης, ανανέωσε την ε, έκκληση που είχε κάνει επανειλημμένα τον τελευταίο καιρό, έτσι ώστε να υπάρχουν συγκλίνουσες ε, δημοσιονομικές ε, πολιτικές, οι οποίες θα εστιάζονται στους οικονομικούς και νομισματικούς στόχους. Πρόκειται για Επομένως, μάλλον πρέπει να δούμε εάν ε, ε, οι οικονομικές πολιτικές των χωρών και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μπορούν να ανταποκριθούν στην έκκληση ε, η οποία τους αποφύθηκε γιατί δεν είναι δυνατόν ένας φορέας μόνος του ή ένα στοιχείο μόνο του να μπορέσει να οδηγήσει σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ούτε θα δώσει την δυνατότητα να γίνουν επενδύσεις τέτοιες που να μπορέσουν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Θα πρέπει να υπάρξει αρκετή ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι κανόνες. Αλλά, από ό,τι φαίνεται, ε, η συζήτηση για τις κυρώσεις για την Ισπανία και την Πορτογαλία, ενώ έχουν κάνει ήδη πολύ μεγάλες προσπάθειες ε, και ενώ η Πορτογαλία για φέτος έχει έλλειμμα χαμηλότερο από το 3%, ε, αυτή η στάση, λέω, έρχεται σε κατάφορη διαφοροποίηση από τα όσα ανα, ε, αναγγέλλονται. Επίσης, με ποιο τρόπο το ευρωπαϊκό εξάμεινο ε, μπορεί να ενδυναμώσει και ενδυναμώνει τις οικονομίες. Θα πρέπει να εφαρμοστεί με τρόπο τέτοιο ε, που να δημιουργήσει πολιτική ευνοϊκή για την ανάπτυξη. μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα και μπορούμε να κάνουμε και καλύτερα. Η, πολιτική η επενδυτική πολιτική ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη θα πρέπει ε, να αλλάξει έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις ασυμμετρίες που αναφέρθηκαν προηγουμένως, ασυμμετρίες ανάμεσα ε, στην Γερμανία, ας πούμε την Ολλανδία και τις χώρες της Ιβηρικής Κερσονήσου ή της Μεσογείου. προβλέπονται όμως αυτά τα μέτρα τα οποία θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε τις ασυμμετρίες ή αντιθέτως τα μέτρα τα οποία προτείνονται ε, θα βαθύνουν και θα ενδύνουν ακόμα περισσότερο τις ανισορροπίες θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια σοβαρή αξιολόγηση των όσων έχουν γίνει μέχρι τώρα και θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική η οποία να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών. Ε, για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει ε, να τροποποιηθεί το ισχύον παρόν πλαίσιο. Σα Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ε, έχω άλλους που επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Κατόπιν τούτου θα κάνω εγώ ένα σχόλιο, γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτά που είπε ο συνάδελφός μου, κύριος Σταρμπάτη, με, μου έδωσε ένα κίνητρο να τοποθετηθώ. Αλλά και από τη συζήτηση ε, ετέθη το ερώτημα γιατί δεν αναπτυσσόμετα επαρκώς. Υπάρχει το θέμα της, του συμφώνου σταθερότητας. Η νομισματική ένεση ε, προφανώς και απαιτεί κανόνες αλλά θα ήμουν πολύ προσεκτικός στο να ισχυριστώ ότι οι κανόνες μας ε, δεν λειτουργούν για τη μείωση του ελλείμματος. Και ο πρόεδρος κύριος Γιούγκερ ισχυρίζεται ότι αν δει κανείς τους αριθμούς, το έλλειμμα της Ευρωζώνης από 6,3 το 2009 έπεσε στο 1,9 το 2016. Δηλαδή πολύ σημαντική μείωση του ελλείμματος. Ω εκ τούτου είναι πολύ δύσκολο να πει κανεί ότι δεν αποδίδουν οι κανόνε Μα αποδίδουν. Σε λίγα μόνο χρόνια μειώσαμε το έλλειμμα, το συνολικό, κατά ένα τρίτο. Ε, Στι ΗΠΑ το έλλειμμα είναι στο 4,4, στην Ευρωζώνη 1,9. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η λύση του προβλήματο είναι να καταργήσει κανεί μόνο το έλλειμμα. Αυτό από μόνο του δεν δουλεύει. Αλλά είναι και δύσκολο να αμφισβητήσει κανεί την άποψη εκείνων ε, που ισχυρίζονται ότι αυτή τη στιγμή έχουμε επιτέλους μία επεκτατική δημοσιονομική πολιτική το 2016, μετά από μία ουδέτερη το 2015, τι θα κάνουμε το 2017. Ε, χρειαζόμαστε να επανέλθουμε προς τα πίσω ή πρέπει να διατηρήσουμε ε, αυτή την ελαφρώς επεκτατική πολιτική του 2016. Εγώ νομίζω ότι η απάντηση είναι απόλυτα σαφής, ότι χρειαζόμαστε ε, το 2017 μία επεκτατική πολιτική και να μην επανέλθουμε σε ε, συρρήκνωση είδαμε ότι το 2009 υπήρχε ε, η ε, ανεπαρκή συνολική ζήτηση. Βεβαίως όλα αυτά δεν αρκούν από μόνα τους. Πρέπει, όπως είπε και ο κύριος Ντράγκη εξάλλου, να έχουμε κατά νου και το θέμα της ποιότητας. Οι επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και ξέρουμε ότι δεν αρκεί η σφαιρική, η συνολική ζήτηση για να υπάρξει ανάπτυξη. Είναι λοιπόν δύσκολο να αρνηθεί κανείς ότι υπάρχει ε, μία κακή σχέση ανάμεσα σε επενδύσεις και αποταμίευση καθόμαστε πάνω σε, έχουμε πάρα πολλά μετρητά, βουνά μετρητών που ε, είτε βγαίνουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε ε, μένουν σε επενδύσεις στις τράπεζες, δεν γίνονται επενδύσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι η στήριξη της ε, δημοσιονομικής πολιτικής είναι το ζητούμενο. Και για μένα είναι δύσκολο να είμαι κατά της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής της ε, ΕΚΤ, κατά της αύξησης της εσωτερικής ζήτησης, κατά του να υπάρχει μία ένωση ε, που να μεταφέρει χρήματα σε εκείνους που τα χρειάζονται κατά του δανεισμού ε, κάτι πρέπει να κάνουμε αν δεν κάνουμε τίποτα πια από όλα αυτά ε, για μένα είναι δύσκολο να δείξουμε και το θέμα μα τελικά πώς θα επιβιώσουμε με αυτό το κοινό νόμισμα θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα Πρέπει να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας και βεβαίω υποστηρίζω ανεπιφύλακτα όλους εκείνους που λένε ότι πρέπει να στηρίξουμε τη σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα, να υπάρχει καλύτερο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών, έτσι ώστε να προκύψουν διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις. Ε, οφείλουμε να εμβαθύνουμε την κοινή αγορά. Αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Εξακολουθούμε να έχουμε χρόνο στη διάθεσή μα. Δεν θέλω να εξάγω τα συμπεράσματα. Αν κάποιο επιθυμεί να λάβει και πάλι το λόγο, ε, πριν δώσουμε το λόγο στον εισηγητή, παρακαλώ μπορεί να τον λάβει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που αναφέρατε ξανά κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια βασικά πράγματα της οικονομικής επιστήμης, αυτά τα οποία έλεγε ο Τζον Μέινταρ Keynes. Αυτό το οποίο έχουμε λοιπόν θα το έλεγε beggar my neighbor policy, δηλαδή προσπαθούμε να αλλάξουμε τις ε, ισοτιμίες. Ε, τι κάνει λοιπόν η Γερμανία, εξάγει αγαθά και εισάγει απασχόληση. Άλλες χώρες στο Νότο ε, εξάγουν απασχόληση και εισάγουν αγαθά, εξάγουν εργαζόμενους. Ο ένα καταστρέφει τον άλλον δηλαδή. Δεύτερον, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε με την νομισματική πολιτική την ε, έλλειψη των επενδύσεων. Μπορεί δηλαδή να γεμίσει με ρευστότητα ε, τη γούρνα εντό εισαγωγικών ο κύριος Δράγκη αλλά πρέπει να φαίνεται και τα άλογα να πιούν. Δεν μπορεί να τα αναγκάσει ο κύριος Δράγκη. Υπάρχουν λοιπόν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες συνεχώς αναβάλλονται γιατί είναι πιο καλό και πιο εύκολο βεβαίως να χρεωνόμαστε με μηδενικά επιτόκια από το να κάνουμε την οποιαδήποτε μεταρρυθμίση. Αυτό είναι το βασικό και βεβαίως ε, μακροπρόθεσμα ε, το τι σημαίνει αυτή η πολιτική αρνητικών επιτοκίων ε, και για τον τραπεζικό τομέα θα είναι καταστροφική. Και το βλέπετε αυτό. Και στη Γερμανία. Και έχουμε, βλέπετε, μία ανακατανομή από κάτω προς τα πάνω. Αν δείτε τις τιμές ε, διαφόρων ε, περισσεκών ε, στοιχείων, ακίνητα, Εργατέχνης. οτιδήποτε. Έχουμε αυτή την ψεύτικη, θα έλεγα, κάλπικη εξέλιξη. Και σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να τα ξαναπώ, να πω ξεκάθαρα το τι πρέπει να γίνει. Εγώ λοιπόν είμαι υπέρ και πρέπει να φροντίσουμε να παραμείνει ενωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν μπορούμε σε βάθος χρόνου να διατηρούμε μια νομισματική ένωση η οποία συνεχώς πηγαίνει να σκάσει. Το σημαντικότερο ερώτημα το οποίο πρέπει να θέσουμε είναι τι είναι αναγκαίο έτσι ώστε να βοηθήσουμε τις χώρες με μεγάλο χρέος πώς θα αποκτήσουν ένα μοντέλο αποδοτικό Πώ θα μπορέσουν να δημιουργήσουν θέσει εργασία στη χώρα τους. Ε, και εντάξει, δεν είναι το θέμα μόνο η Ελλάδα, είναι το θέμα των ε, χρημάτων που έχουν οι τράπεζε στην Ελλάδα. Τα χρήματα αυτά ξαναραίουν στην χώρα. Λοιπόν, και ε, θα, θα σταματήσω κύριε Πρόεδρε. Μπορούμε να βοηθήσουμε λοιπόν την Ελλάδα ως εξής βρείτε μία ισοτιμία συναλλαγματική που θα σας κάνει ανταγωνιστικούς. Αυτή είναι η δυνατότητα και έτσι θα αντικαταστήσετε την ε, κατανάλωση παραγωγή. Πραγματικά σας λέω αγαπάω την χώρα, δεν θα πιστέψετε με ένα ανταγωνιστικό νόμισμα και πόσοι τουρίστες θα έρθουν στη χώρα. Και αυτό το οποίο χρειάζεται λοιπόν η χώρα είναι και μία διαγραφή του χρέους δεν θα μπορέσει ποτέ να το πληρώσει ποτέ. Γι' αυτό ζητάω λοιπόν να της δώσουμε και μια άφεση χρέους αν θέλετε. Και όλοι γνωρίζουν σε αυτή την αίθουσα πως ένας επιχειρηματίας ο οποίος χρεοκοπεί πρέπει να έχει την δυνατότητα να ξαναδραστηριοποιηθεί και χρειάζεται ακριβώς ένα πρόξιμο να πάρει ε, Αυτά τα τρία χρειαζόμαστε λοιπόν όπως σας είπα. Νέα συναλλαγματική ισοτιμία και ε, διαγραφή χρέους και μια νέα όθηση. Αλλά να περιμένουμε να βρέξει μάνα εξ ουρανού δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου ξαναδώσετε το λόγο. Thank you very much. Εγώ σας ευχαριστώ. Γίνεται ζωντανή η συζήτηση. Πολύ ωραία. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά στη διάθεσή μας. Βλέπω τον συνάδελφο από τις κάτω χώρες πρώτα. και μετά ο Σάνσος Περέιρα. Έντονη η συζήτηση και μου αρέσει. Λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξή. Εγώ είμαι εδώ γιατί θέλω να διατηρηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη χώρα μου υπάρχουν κόμματα που θέλουν να καταρρεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί θέλουμε να παραμείνει ενωμένη και ισχυρή. Οπότε ο συνάδελ, η συνάδελφος από την Πορτογαλία είπε ότι ε, αν τιμωρηθεί η Πορτογαλία θα μειωθεί η στήριξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη χώρα μου σημαίνει το αντίστροφο. Αν υπάρχουν κανόνες και δεν τηρούνται και δεν τιμωρηθεί όπω λέτε η Πορτογαλία, θα μειωθεί η στήριξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη δική μου χώρα. Τι είναι λοιπόν η συζήτηση. Υπάρχει και η Ισπανία. Η συνάδελφο είπε ότι η Γερμανία και η Ολλανδία έχουν πλεόνασμα. Ε, μα, ναι, είμαστε υπερήφανοι. Μεταρρυθμίσαμε την οικονομία μα. Χτες ακούσαμε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ πώ είμαστε η τέταρτη χώρα, αν δείτε την ανταγωνιστικότητα. μα μας ικανοποιεί αυτό και μεταρρυθμίσαμε και κερδίσαμε εκλογέ με αυτό το πρόγραμμα. Ε, οπότε ε, δεν θα γίνει κανείς ισχυρότερο μέλος τη Ευρωπαϊκή Ένωση με το να ξασθενήσουν τα ισχυρότερα μέλη. Αυτό θα ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, το ζήτημα είναι ε, να κάνει κανείς ε, το σωστό και επομένως οι κανόνες να είναι ευφυείς και σωστοί. Ενδεχομένως ίσως έχουμε διαφορετική ε, ιδέα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν έλλειμμα κάτω από το 3% αλλά εάν δεν υπάρξει αρκετή ανάπτυξη τότε υπάρχει μια, μπορεί να υπάρξει μια απόφαση για μείωση των διαφορετικών ταμείων αλλά το θέμα είναι από ποια πλευρά το λούς θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι ευφυές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ο κύριος από την Πορτογαλία. Είναι καλό που ανάβουν λίγο τα αίματα και χαίρομαι ως οικονομολόγος γιατί με ενδιαφέρει πολύ αυτή η συζήτηση. Ε, σχετικά με τα όσα ε, είπε προηγουμένως ε, ο κύριος Σερβατή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι δεν ε, έχουμε και τίποτα άλλο να κάνουμε όσον αφορά ε, την οικονομική πολιτική. Ξέρουμε ότι ε, τα κόκκινα δάνεια είναι μεγάλη τροχοπέδη. Και επομένω επικεντρωνόμαστε στην δημοσιονομική πολιτική. Όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική, εγώ θα ήθελα να θέσω ένα κεντρικό επιχείρημα. Έχω εδώ τον αγαπητό συνάδελφο από την Ολλανδία, ο οποίος τεκμέρι ότι οι μακροοικονομικές ε, ανισότητες που υπάρχουν σε ορισμένε χώρες, ας πούμε, ευθύνονται, ε, ε, μάλλον για αυτά ευθύνονται αποκλειστικά οι χώρες. Εγώ όμως λέω ότι είναι μοιρασμένη η ευθύνη. Ε, είναι όντως υπάρχουν χώρες οι οποίες έκανε κάποιες έκακες πολιτικές στο παρελθόν, αλλά έχουν πλέον και αυξημένα προβλήματα και φτώχεια και λόγω ακριβώς των πολιτικών λιτότητας. Και αυτό το υπενθυμίζουν άλλωστε ε, και οι εκθέσει των πέντε προέδρων. Ρωτώ τους συναδέλφους, ε, ξέρετε κάποια νομισματική περιοχή ε, που να μην έχει δημοσιονομική ενότητα, να μην έχει δηλαδή ενιαία δημοσιονομική πολιτική. Δεν είναι δυνατόν, εάν δεν έχουμε ενιαία δημοσιονομική πολιτική, να, να δημιουργήσουμε έναν καλά ενωμένο νομισματικό χώρο. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν αυτή η Fiscal Union ε, θα πρέπει να ε, έχουμε βελτίωση σε όλες τις χώρες, ε, αλλά εάν συνεχίσουμε, όπως λένε ορισμένοι ακραίοι, ότι η Ελλάδα και η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν και μακροοικονομική ανισότητα και ευθύνονται αποκλειστικά αυτές και εδώ να πω εν παρόδο ότι και η Γερμανία έχει, ένα, έχει MIP αλλά εν πάση περιπτώσει ε, ας μην το συζητήσουμε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες ε, όπως η Πορτογαλία ας πούμε θα συνεχίσουν ε, με την εξυγίανση των πολιτικών τους αλλά η Γερμανία και κάποιες άλλες χώρες οι οποίες ε, ενδεχομένως πάνε καλύτερα θα πρέπει να διευρύνουν τη φορολογική τους πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Ο Έλληνας συνάδελφος, ο κ. Μπαλάουρος, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πράγματι ο διάλογος ε, άναψε. Ε, μία παρατήρηση για τα κράτη όπως η Ολλανδία. Θα πρέπει, συνάδελφε, να έχουμε υπόψη μας και την ιστορικότητα. Δηλαδή τα τελευταία 50-60 χρόνια τι πέρασε κάθε χώρα, τι καταστροφές, τι επεμβάσεις έγιναν ε, και το πιο παλιό παρελθόν αν ήταν απεικιοκρατική δύναμη ή οτιδήποτε άλλο και έφτιαξε πρωτογενή πλούτο και πορεύτηκε στην πορεία. Αλλά είναι μια άλλη ιστορία αυτή να πούμε για τα ιστορικά δεδομένα. Τώρα, ε, είπε κάποιος συνάδελφος για, για το Brexit ότι καλύτερα είναι να πάμε στο εθνικό νόμισμα και ακόμα και με, καλή ε, ισοτιμία μια παρατήρηση εδώ, η ισοτιμία που μπήκαμε, όχι μόνο η Ελλάδα στο ευρώ, αλλά και πολλά άλλα κράτη, νομίζω και είχε αποδειχτεί εκ των υστέρων ότι ήταν δυσμενής για τις χώρες αυτές. Κυριάρχησε το Μάρκο και η ισοτιμία ήταν δυσμενής. Τώρα, ε, να σας πω, η Ελλάδα είναι σε πρόγραμμα έξι χρόνια. 6 χρόνια. Έτσι. Τι είχαμε σαν συνέπεια, προσέξτε το καλά και μετά λιδωρίστε τους Έλληνες ή την Ελλάδα. Το χρέος. Το χρέος υπερδιπλασιάστηκε. Υποτίθεται ότι πήγαμε σε πρόγραμμα για να μειώσουμε το χρέος. Υπερδιπλασιάστηκε. Η ύφεση, η ύφεση έφτασε 25%. Ούτε στο μεγάλο κράκ της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είχαμε 25% ύφεση. Η ανεργία έφτασε 27% εκ των οποίων οι νέοι μας, μας άνθρωποι επιστήμονες και πολύ καλοί επιστήμονες είναι 60% άνεργοι και έχουν πάει και, και αιμοδοτούν τα μεγάλα κράτη της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αυστραλίας έτοιμοι επιστήμονες, γιατροί, μηχανικοί από ε, ε, ε, με το αίμα του, του απλού Έλληνα που τους σπουδάσαμε έχουν φύγει και έχουν πάει σε αυτές τις χώρες. Το δούνου του μετά από το, το, διεθνές, το Διεθνές Νοσηματικό Ταμείο μετά από τέσσερα χρόνια είπε ότι έκανα λάθος στους πολλαπλασιαστές και το πρόγραμμα βγήκε έξω. Έκανα λάθος τώρα μιλάει για τις συνέπειες των κοινωνικών επιπτώσεων στη χώρα όταν το 33% του ελληνικού λαού είναι σε απόλυτη φτώχεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχουμε επίσης και τώρα δεν μπορούμε να κυβερνήσουμε. Είμαστε σε επιτήρηση όχι μόνο στα οικονομικά δεδομένα αλλά ακόμα και για την παιδεία το τι διδασκαλία θα κάνουμε στην παιδεία παρεμβαίνουν ή παρεμβαίνει η Τρόικα. Α, περί αυτού πρόκειται. Δεν έχετε καταλάβει μάλλον. Δεν αφορά μόνο την οικονομία. Και έχουμε για την οικονομία να πούμε και μερικά άλλα πράγματα που είμαστε επίσης επιτήρηση και για πολλά άλλα. Είναι ότι ε, θέλουν πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% κάθε χρόνο. Ποια, ποιο κράτος, ιστορικά, ιστορικά, ποιο κράτος, εσείς μιλάτε τώρα για έλλειμμα το 3% ή το 2,5% και κτλ. Άκουσα κάποιους συναδέρφους. Ιστορικά ποιο κράτος μπορεί να βγάλει 3,5% κάθε χρόνο πλεόνασμα για να το δίνει στη, στους πιστωτές μας. Σε βάρος της ανάπτυξης. Σε βάρος της ανάπτυξης. Και τελευταίο πράγμα, το χρέος το χρέος, σας είπα προηγουμένως, υπερδιπλασιάστηκε με τη συνταγή της Τρόικας κτλ. Ωραία. Μπορεί να, να απομειωθεί. δεν θέλω να επιχειρηματίσω πολύ γι' αυτό, είπαν και άλλοι συνάδελφοι, νομίζω ότι έχουν δίκιο, θα φανεί αυτό, θα φανεί, δεν μπορεί μια χώρα η οικογένεια ή η επιχείρηση με ένα κρέο τέτοιο να, μπορέσει να, να προχωρήσει. Just to be, because a lot of colleagues and we have few minutes. Yeah, yeah, uh, uh, Just a moment, please. Just a moment. Ε, ε, επομένως ζητάμε απομείωση του χρέους. Έτσι. Θυμίζω το ιστορικό προηγούμενο ότι η Ελλάδα μαζί με άλλα κράτη, η φτωχή Ελλάδα μετά τον πόλεμο το 1953 συνέβαλε στην απομείωση του χρέους της Γερμανίας. Η Ελλάδα, το θυμίζω αυτό για τους φίλους μας, όχι μόνο τους Γερμανούς, από όλου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Thank you. Could you please try to one... Λοιπόν, αν έχει την καλοσύνη, ένα με δύο λεπτά ο καθένας για να μπορούν να μιλήσουν και άλλοι. Κοιτάξτε, εδώ προσπαθούμε να βρούμε καλές πολιτικές. Αλλά τι να σας πω, αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για το τι γίνεται, τι να πω κι εγώ. Πραγματικά εντυπωσιάζομαι ακούγοντας ε, ότι το, η ποσοτική χαλάρωση είναι εκείνη η οποία προκαλεί χαμηλά αρνητικά επιτόκια. Το αντίθετο συμβαίνει. Η ποσοτική χαλάρωση είναι το αποτέλεσμα της ε, μείωσης ε, των επιτοκίων. Τι νόημα έχει να αξιολογεί κανείς τα αρνητικά επιτόκια. Το νόημα είναι να ε, μπορεί κανείς να εξοικονομήσει επενδύσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο. Αυτά που σας πω είναι βασικά θέματα της μακροοικονομίας. Είναι βασικές αρχές. Τώρα το να επικρίνει κανείς την ποσοτική χαλάρωση ε, δεν μπορεί να την ε, σχολιάζει ως καθοριστικό παράγοντα. Δεύτερον, η ποσοτική χαλάρωση είναι σαφές ότι δεν αρκεί για να στηρίξει τη ζήτηση και την οικονομική ανάπτυξη και κατ' ουσίαν συζητάμε το πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε την ε, ε, νομισματική πολιτική μέσα από τη δημοσιονομική πολιτική και τις επενδύσεις πολύ καθοριστικά αυτά για να ε, αναζητηθεί ε, μια καλή θεραπεία και ε, μια καλή συνταγή. Και τέλος, όταν λέτε ότι η ποσοτική χαλάρωση μειώνει το ποσοστό των μεταρρυθμίσεων, τι να πω κι εγώ τώρα. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Και εγώ μπορώ να πω ότι υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες προχωρούν σε περισσότερες μεταρρυθμίσεις και άλλες σε λιγότερες. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι να έχουμε ένα επεκτατικό μακροοικονομικό πλαίσιο. Είναι πολύ σημαντικό να ε, μπορεί κανείς να τα ιεραρχεί τα πράγματα, αν τα ανακατεύει όλα. Ε, είναι πολύ δύσκολο να εξευρεθούν λύσεις. Silva Pereira. Uh, thank you, Κοιτάξτε, όσον αφορά την κατάσταση στην ε, Πορτογαλία, όπως είπε και ο συνάδελφος, η Πορτογαλία για τρία χρόνια πέρασε μέσα από ένα δύσκολο πρόγραμμα προσαρμογής. Και αυτό το σχεδίασαν ευρωπαϊκοί θεσμοί αυτό που δεν θα καταλάβουν ποτέ οι άνθρωποι στην Πορτογαλία είναι ότι στο τέλος ενός τέτοιου σκληρού προγράμματος όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθούσε όλες τις εξελίξεις αν θέλετε, ξέρετε, μπορώ να σας φέρω και να σας δείξω ε, τόμους ε, ε δηλώσεων όπου συνέχεραν την ε, πορτογαλική οικονομία γιατί ε, σε τελική ανάλυση το 2015 είχαν, ε, είχαμε πετύχει τους στόχους μας, αλλά παρόλα αυτά θα μας επιβάλλουν κυρώσεις. Η ίδια Επιτροπή βέβαια που μας συνέχερε. Αυτό δεν βγάζει κάπου νόημα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ο Ολλανδός συνάδελφος μοιάζει να πιστεύει ότι υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι αν δεν ε, εφαρμόζει κανείς ε, τους στόχους θα πρέπει να τιμωρείται. Εγώ πρέπει να σας ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει αυτό στην ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Έχουμε το άρθρο 23 παράγραφος 11 που λέει με απόλυτη σαφήνεια ότι αν δεν επιτυγχάνεται ο στόχος λαμβάνεται μία απόφαση και η απόφαση αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη της όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αυτές που θα δώσει και φέτος η Πορτογαλία για να πετύχει το στόχο του 3%. Βεβαίως και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της αναλογικότητας, όπως επίσης ε, και ε, το τι γίνεται στην πραγματική οικονομία. Αυτό είναι ο κανόνα. Αν κάποιο τώρα στην Ολλανδία ερμηνεύει διαφορετικά τους κανόνες, νομίζω ότι οι πολιτικοί θα πρέπει να εξηγήσουν στου πολίτες τι ακριβώς λένε οι κανόνε. Thank you. Uh,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 κάποιες ε, κατευθύνσεις και ανταυτού αυτό το οποίο άκουσα ήταν παρά, ε, παράπονα και γκρίνια. Δεν ε, είδα καμία αποφασιστικότητα. Δεν άκουσα κάποιον να πει ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τη δική μας χώρα. Έτσι με με περισσότερη ειλικρίνεια. Δηλαδή, αν πρέπει να παραπονιέται κανεί, πρέπει να παραπονιόμαστε εμεί από τη Βουλγαρία. Γιατί επί σειρά ετών ήμασταν πολύ αυστηροί στη δημοσιονομική πειθαρχία. Επίση, τα σύνορα τη Βουλγαρία είναι εξωτερικά σύνορα. Ε, προσπαθούμε κάπως να ανταποκριθούμε στην τεράστια μεταναστευτική πίεση και λόγω αυτού η Ευρώπη δεν έχει πλημμυρίσει εντελώς από μετανάστες. Η Βουλγαρία είναι φτωχή χώρα. Πάνω από 2 εκατομμύρια Βουλγαροί ζουν με 150 ευρώ το μήνα. Το μήνα, όχι τη μέρα. Και όπως οι περισσότερες χώρες που συζητάμε εδώ πέρα, μέχρι προσφάτως η Ελλάδα απειλούσε τους πολίτες τους και τους έλεγε θα βουλγαροποιηθείτε. Θα γίνουν σαν Βούλγαρη. Κι όμως είπε οι Έλληνες βγαίνουν στη σύνταξη με 700 ευρώ ελάχιστη σύνταξη. Στη Βουλγαρία είναι 75 ευρώ η ελάχιστη σύνταξη. Γι' αυτό όταν μίλησα πριν είπα ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η εμπιστοσύνη. Η Βουλγαρία είναι όπως σας ε, περιέγραψα. Η Ευρώπη απ' την άλλη δεν θα πρέπει να είναι κατακαιρματισμένη γιατί αν αποσυνδεθεί θα επιστρέψουμε στον 17ο ή 18ο αιώνα. Αυτό θέμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε τόσοι έξυπνοι άνθρωποι στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό λοιπόν να διαχειριστούμε πράγματι τις ε, χρηματικές ροές γιατί οι τράπεζες έχουν μετρητά, χρειαζόμαστε επενδύσεις και όμως κανένας δεν μιλάει πώς θα γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, είδα τον κατάλογο των μιλητών και θα δώσω τον λόγο γρήγορα στον εισηγητή γιατί θα ε, επισκεφτεί το Κοινοβούλιο Διοικητή τη Τράπεζα τη Γαλλία και πρέπει να πάω να τον υποδεχτώ. Κύριε Σάντι, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πω ήταν μια έντονη, ενδιαφέρουσα συζήτηση. Παραγωγική και για εμένα ε, ως εισηγητή Πολλές ε, από αυτές τις ιδέες ε, βεβαίως έχουν ακουστεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι ιδέες του κυρίου Σταρμπάτη ε, τις οποίες αντιλαμβάνομαι να σας πω σε προσωπική βάση. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Η Ευρωζώνη δεν είναι ιδανική νομισματική ζώνη. Οπότε τι κάνουμε. Διαχειριζόμαστε διαδικασίες οι οποίες δεν είναι οι βέλτιστες. Γι' αυτό ακριβώς δεν βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα τα οποία θα ανταποκρίνονταν στην εντολή και στο χρονοδιάγραμμα του Κοινοβουλίου. Αλλά πέρα από αυτό το πραγματικό πρόβλημα που πρέπει να δούμε, πέρα από τις συστάσεις αναχώρα, είναι το εξή. Δεν συμβαίνει οικονομική σύγκληση. Υπάρχει οικονομική απόκληση και οι πολιτικές τις οποίες συζητάμε δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Μιλάμε για σύγκληση πολιτικών όσον αφορά πίνακες βαθμολογίας που έχουμε, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε το πραγματικό πρόβλημα της σύγκλησης του βιωτικού επίπεδου, της οικονομικής παραγωγής, κατά κεφαλήν. Και αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου του ότι οδηγούμε, λειτουργούμε όπως σας είπα με συνθήκες ε, και με όρια νομισματικής ζώνης τα οποία δεν είναι ιδανικά ο κύριος Σταρμπάτη δεν το αποδέχεται λέει 3 και 3 κάνουν 6 αλλά στην πραγματικότητα και έχει δίκιο σε αυτό αλλά έχουμε ένα πολιτικό κατασκεύασμα το οποίο δεν είναι βέλτιστο από οικονομική και χρηματοπιστωτική πλευρά πρέπει με αυτό τι πολιτικές να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Στο παρελθόν με αυτές τις μη βέλτιστε συνθήκε είχαμε πετύχει καλύτερη απασχόληση και περισσότερες επενδύσεις. Παρόλο το πλαίσιο, νομίζω λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στα επίπεδα εκείνα τα οποία ήταν πάρα πολύ καλά σε σχέση με το που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ και εγώ. Νομίζω λοιπόν πως η συζήτηση μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων ε, είναι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο είναι ένας όρος για να προχωρήσουμε και να μην είμαστε έτσι, λιγότερο από βέλτιστοι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. 11 Οκτωβρίου για την έκθεση θα εξετάσουμε τις τροπολογίες και θα ψηφιστεί στην Επιτροπή και δύο... στη δεύτερη οκτω... Ολομέλεια του Οκτωβρίου θα πάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ ιδιαίτερα και τους βουλευτές από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, επόμενη συνεδρίαση Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, ακριβώς το θέμα οικονομικός διάλογος για Πορτοκαλία και Ισπανία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.